Euh, euh, Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Προς το παρόν να κολλείται η Πρόεδρος. Ε, ότι έχουν κρατήσει κάποιες διαδηλώσεις για τους σιδηροδρόμους. Ε, δεν ξέρω αν θα παραμείνει όμοιρος σε αυτό το αυθόρμητο κίνημα που δημιουργήθηκε. Προς το παρόν θα προεδρεύσω εγώ λοιπόν. Καταρχήν να εγκρίνουμε την σε διάταξη αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Επίσης, να εγκρίνουμε τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων. Και μια και απουσιάζουν αρκετοί συντονιστές γιατί είναι στη Λιουμπλιάνα. Φαντάζομαι μερικοί θα πάτε από το απόγευμα ή αύριο. Αναβάλλεται η συνεδρίαση των συντονιστών που είχε προγραμματιστεί για σήμερα. Οπότε, κανονικά θα διακόψουμε το μεσημέρι στις 11.30 και θα ξαναρχίσουμε στις 2.30. Οπότε έχουμε λίγο χρόνο, αλλά ελπίζω να είμαστε αποτελεσματικοί. Ε, αν δεν έχετε αντίρρηση θα περάσουμε κατευθείαν στις ψηφοφορίες. Θα κάνουμε όμως πρώτα μία δοκιμή για να εξετάσουμε την απαρτία και να ξεκριβώσουμε τους ψήφους των ομάδων. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, κάποιος συνάδελφος δεν έχει την κάρτα, οπότε θα σηκώνει χέρι. Καλώς. το σύστημα λειτουργεί και μια και το ΕΡΚ δεν έχει υπεράριθμους, όλα καλά. Ο κύριος Νταλούντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά την ε, έκθεση τα παρντέλ, ε, ενώ δεν γνωρίζω το περιεχόμενο, ήθελα να πω ότι λάβαμε πολύ αργά τα έγγραφα για να εξετάσουμε. Ε, οπότε δεν θέλουμε να την ψηφίσουμε ακόμα. Ευχαριστώ. Bien, merci. Euh, là, je pense être... Ευχαριστώ. Εύλογη η παρατήρηση. Κανονικά πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 24 ώρες πριν την, το κατάλογο ψηφοφορίας μετά την οριστικοποίηση. Αλλά έχουμε και εμείς ε, κλονιστεί κάπως από όσα συμβαίνουν και στην Επιτροπή. Η κυρία Ταπαρδέλ θα μιλήσει για την έκθεσή της. Ο κατάλογος της ψηφοφορίας εστάλει χθες. Ε, ε, Πιθανότατα είναι λάθος της γραμματείας ε, και μιλήσαμε με τους πράσινους στο τηλέφωνο και τους είπαμε ότι ε, έχει σταλεί ο κατάλογος της ψηφοφορίας και τους μιλήσαμε μαζί τους χθε το πρωί. Δεν ξέρω τι συνέβη λοιπόν. Αν πάντως ε, έχει γίνει κάποιο λάθος, δεν είναι δικό μου λάθος. Μάλλον σε επίπεδο γραμματείας κάτι συνέβη. <coughs> Κυρία Ταπαρδέλ, κανείς δεν σας κατηγόρησε. Κανένας ε, δεν σας ε, κατηγόρησε. Όχι, δεν το πήρα προσωπικά. Απλώς θέλω να διευκρινίσω ότι ο κατάλογος ψηφοφορίας εστάλει χθε. Κανονικά όλοι έπρεπε να τον είχαν λάβει. Ναι, εντάξει, τον έχουμε λάβει πια τον κατάλογο, οπότε κανένα πρόβλημα ψηφοφορία της πρώτης έκθεσης του κυρίου Ερτούγκ για το πείραγμα των χιλιομετρητών, την παραποίηση των χιλιομετρητών σε μηχανοκίνητα οχήματα. Ξεκινάμε. Ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 46. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. 47. 47, Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 47. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 48. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται. Τροπολογία 49. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 και 51 ήταν μαζί. 52 τώρα. 52. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία συμβαστική 3. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 63. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 64. Υπέρ κατά αποχές θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά συμβαστική τροπολογία 5 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 6 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 77, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 7, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 79, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 80. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 86 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 88 Εδώ έχουμε κατά τμήματα ψηφοφορία. Ζήτησαν οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες. Για το πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος του πρώτου τμήματος της 88 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται το πρώτο τμήμα, οπότε το δεύτερο μάλλον καταπίπτει. Τροπολογία 91. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 92. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 93. Καταπίπτει. Περνάμε στα παραρτήματα. Τροπολογία 96. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ Α, όχι καταπίπτει, όρη συγγνώμη 98 και 99 μαζί ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται τροπολογία 100 και 101 ή μάλλον καταπίπτουν Πάμε στην 103. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 105. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 104 καταπίπτει ή 106 το ίδιο. 107. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 102 καταπίπτει και πάμε στη συμβαστική τροπολογία 9. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 112 και 113 είναι πανομοιότυπες Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 114 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 115 καταπίπτει. 117. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 118 καταπίπτει. Το ίδιο και 119. 120. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 121 καταπίπτει, 122 ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι υπέρ της 122, κατά, αποχές εγκρίνεται, 123 ποιος είναι υπέρ, κατά, 123. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 124 καταπίπτει. Συμβαστική τροπολογία 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 127. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 128. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 8 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 9 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11 γλωσσική τροπολογία. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Συμβαστική τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 13 καταπίπτει. Τροπολογία 15. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 28 και 35 μαζί. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 36. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 37. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 38 και 39 μαζί. Υπέρ είναι το κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 40. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Και πραγματικά πρόκειται για θρίαμβος, 46 ψήφοι υπέρ, μία μονοκατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Περάσουμε, να περάσουμε τώρα στο δεύτερη και τελευταία ψηφοφορία, που είναι η ψηφοφορία της έκθεσης της κυρίας Κλόντια Τσαπαρντέλ για τους κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην κοινότητα. Έτοιμοι για τη δεύτερη ψηφοφορία. Georges. Έτοιμος. Ωραία λοιπόν, ξεκινούμε με τη δεύτερη ψηφοφορία. Τροπολογία 4, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6, πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται κατά την άποψή μου. Να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά επαλήθευση γιατί την συμβιβαστική ε, τροπολογία. Νομίζω όμως ότι απορρίπτεται. Πέρασε τις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται πράγματι. Επομένως, ψηφίζουμε την τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, Νομίζω ότι έχουμε πάλι τις ίδιες πλειοψηφίες. Ε, επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Πράγματι, απορρίπτεται με 25 ψήφους κατά και 23 υπέρ. 6, δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πάλι έχουμε την ίδια πλειοψηφία, απορρίπτεται. Εντάξει, να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τι έγινε? Έχουμε διαμαρτυρίες πέρα της ψηφοφορίας. Πράγματι, πάλι την ίδια πλειοψηφία, 23-25 απορρίπτεται, η τροπολογία 2 αποσύρθηκε, τροπολογία 13. Υπέρ της 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 8 και τροπολογία 9 που είναι ταυτόσιμες ψηφίζουμε μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. Τροπολογία. Ησυχία παρακαλώ. Τροπολογία 10 και 11 ταυτόσιμες πάλι. Ψηφίζουμε μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία 12 12 καταπίπτει. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14 και τροπολογία 3 αποσύρθηκαν. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Έχουμε πάλι την ίδια πλειοψηφία. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να επαληθεύσουμε και πάλι ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Το ΕΛΚ ε, πολύ μιλάει σήμερα. Λαλίστατη. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ησυχία. Να ψηφίσουμε τώρα, ζητώ συγγνώμη, το κείμενο στροποποιήθηκε ηλεκτρονικά βεβαίως, άρχεται η ψηφοφορία. Τελική ψηφοφορία για την έκθεση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 25 ψήφους υπέρ, 22 κατά και μία αποχή. Η κυρία Τσαπαρντέλη ζητά το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι ήταν ε, πολύ δύσκολο αυτό το θέμα και στη διαπραγμάτευση και ε, με τις πολιτικές ομάδες και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ ε, τήρησα ανοιχτή στάση, προσπάθησα να καταλάβω αυτό που μου ζητούσε η Επιτροπή, δηλαδή τι πρόβλημα υπάρχει με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Καλώς, θα μιλήσω αγγλικά, λέμε η Ήταν πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και ευθύ εξ αρχή προσπάθησα να το επιλύσω με το σωστό τρόπο. Συζήτησα με την Επιτροπή και καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι θέλουν να επιλύσουν το πρόβλημα που έχει προκύψει με τις ΗΠΑ. Αλλά νομίζω ότι τα δικαιώματα των επιβατών και τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων είναι πολύ σημαντικά. Διότι εδώ δεν αναφερόμαστε μόνο στι Ηνωμένε Πολιτείε, αναφερόμαστε σε έναν από του πιο σημαντικού κανονισμού για την αεροπορία το 2008 το 2008 του 2008. Ε, είχα διαπραγμάτευση και με τους άλλους και ηγητές και πραγματικά με εκπλήσει το γεγονός ότι παρά το γεγονός ότι υπήρχε συμφωνία με τους αδέλφους από το ΕΛΚ, δεν τήρησαν τη συμφωνία και δεν μπορούν να μου λένε τώρα ότι έχω άδικο, διότι υπάρχουν αποδείξεις, υπάρχουν email που στείλαμε ένα στον άλλον, στα οποία είχαμε συμφωνήσει. Και είχα και τη διάθεση να λύσω το πρόβλημα και να αποσύρω κάποιες από τις τροπολογίες μου που ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Λυπάμαι που τηρούμε μια τέτοια στάση όταν κανονικά θα έπρεπε εδώ να βασιζόμαστε σε δικαιοσύνη και είναι κρίμα που αντιμετωπίζουμε ένα τόσο σημαντικό θέμα με τέτοιο τρόπο. Η πλειοψηφία δεν είναι 26 άτομα στη τελική ψηφοφορία. Θα ήθελα λοιπόν να μην ψηφίσετε την εντολή για το Συμβούλιο, γιατί δεν έχουμε πλειοψηφία 26 ατόμων. Ζητώ λοιπόν να μην ψηφίσουμε την εντολή προς το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις εξηγήσεις σας. Επομένως δεν θα ψηφίσουμε την εντολή. Δεν ψηφίζεται. Με αυτό λοιπόν κλείνουν οι ψηφοφορίες. Ψηφίσαμε τις δύο εκθέσεις και περνάμε στο επόμενο σημείο της σα διάτοξης. Η έκθεση της κυρίας Δανιέλα Γιούτο για τις συνδυασμένες μεταφορές. Επειδή έχουμε συνήθως ε, ε, φασαρία μετά το πέρα τη ψηφοφορία. Θα περιμένουμε δύο λεπτά για να βγείτε η και μετά θα δώσω το λόγο στην κυρία Γιούτο. Κυρία Φώστερ, μήπω να βγουν οι υπόλοιποι. Όχι, συγγνώμη, είναι διαδικαστικό. Στη δική μου τη μετάφραση. Όταν ε, είπαμε για την ψηφοφορία προς το Συμβούλιο, δεν άκουσα πολύ καλά και είπατε θα ψηφίσουμε για το Συμβούλιο, ενώ η συγγήτρια αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο αριθμό ψήφων. Δηλαδή, εάν δεν ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή και δεν έχουμε 26 και παραπάνω ψήφους, δεν μπορούμε να πάμε στον τριμερή διάλογο. Θα μπορούσε κάποιος να μου το διευκρινίσει αυτό. δεν έχω την αίσθηση ότι άλλες πολιτικές ομάδες δεν ήθελαν να πάει το θέμα στο Συμβούλιο. Αυτό θα γίνει αυτή τη φορά. Εγώ δεν κατάλαβα αυτό ακριβώς. Θα πρέπει να ψηφίσουμε, διότι δεν υπάρχει ξεχωριστό άρθρο για τα θέματα αυτά. Αν υπάρχει πλειοψηφία για να ε, υπάρξει τριμερής διάλογος, υπάρχει πλειοψηφία και πρέπει να το ψηφίσουμε. Ο Πρόεδρος. Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος κανόνας για το πώς πρέπει να ψηφίζεται μια εντολή και να γίνονται πόρους και να λέμε ότι μετά από την ψηφοφορία της έκθεσης ε, πρέπει να ψηφίσουμε και για την εντολή. Το θέμα είναι ότι η συγκήτρια έδωσε κάποιες εξηγήσει και θεωρεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ε, και ότι οι συντονιστές ε, δεν είναι σε θέση να το αποφασίσουν. Μετά από τη συνάντηση των συντονιστών θα προτείνουμε να ψηφιστεί μετά την, ε, στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής. Είναι απλώς μια καθυστέρηση, αλλά δεν ε, υπάρχει κάποιο άρθρο το οποίο να λέει ότι λόγω του αριθμού των ψήφων πρέπει να γίνει ή δεν πρέπει να γίνει ψηφοφορία. Ναι, αλλά όσο έχει αυτή τη στιγμή, εντάξει, με την επιφύλαξη του γεγονότο ότι δεν είναι παρόντε οι συντονιστέ, τέλο πάντων δεν μα ενδιαφέρει. Εμεί είμαστε ε, μια επιτροπή η οποία μπορεί να αποφασίσει. Καταλαβαίνω την απογοήτευση και την ενόχληση της εισηγήτριας. Δεν είναι προσωπικό το θέμα βεβαίω, αλλά το θέμα είναι ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που είναι εδώ στις ομάδες ε, καταψήφισαν την έκθεση. Εάν λοιπόν ε, ε, αυτομάτως το θέμα πάει στην Ολομέλεια, θα είναι εκεί όλες οι πολιτικές ομάδες και θα γίνει ακριβώς το ίδιο. Για μένα ουσιαστικά είναι χάσιμο χρόνο αυτό. Το καλύτερο είναι να ψηφίσουμε για να δούμε αν θα πάει στον τριμερή διάλογο, διότι εδώ θα έχουμε την Επιτροπή, το Συμβούλιο και την Εισηγήτρια και θα μπορούν να προχωρήσουν οι συζητήσεις. Πριν χρειαστεί να πάει στην Ολομέλεια. Σε εσάς, από εσά εξαρτάται, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί να πρέπει να ακολουθήσουμε διαφορετική διαδικασία και να μην ψηφίσουμε τώρα για να ξεκινήσει η εντολή, ε, όπως και σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό απλώς ήθελα να πω. un petit euh. Υπάρχει, κυρία Φώστερ, ένα προβληματάκι. Θα τα πω λίγο ήρεμα. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Κάποιοι φύγανε στο μεταξύ. Δεν είμαι βέβαιος ε, ότι αν ψηφίσουμε τώρα θα έχουμε ακριβώς ε, την ίδια πλειοψηφία και ε, το ίδιο αποτέλεσμα ουσιαστικά. Προτείνω λοιπόν ότι ακόμα και αν υπάρχει συμφωνία, θα ήταν ίσως καλύτερα να ψηφίσουμε για την εντολή στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής και μετά να το έχουμε συζητήσει και με τους κοιόδης και με τους συντονιστές ε, και να γίνει ψηφοφορία. Διότι κάποιοι έφυγαν και θα αλλάξει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Ζητώ συγγνώμη, δεν ε, ήμουν αρκετά γρήγορος ίσως, δεν σας έδωσα καιρό το λόγο. Έγιναν πολύ γρήγορα τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι αλλάζει τίποτα επί της ουσίας. Θα υπάρχει η ίδια πλειοψηφία νομίζω. Πρέπει να υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία της Επιτροπής. Πιανού το τηλέφωνο του κυρίου Κόχ μάλλον. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία θα σας δώσω το λόγο, ναι, μην ανησυχείτε, αλλά νομίζω το πιο λογικό είναι να αναβάλουμε. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ο Άντερσον. Κύριε Πρόεδρε, δεν νομίζω ότι κάνετε κάτι λάθο και η κυρία Φώστερ κάνει λάθο. Γιατί το άρθρο 69C λέει σαφέστατα ότι η Επιτροπή μπορεί, έχει ένα μέι δυνητικό, δεν έχει σάλ υποχρεωτικό. Η κυρία Φώστερ καλό θα ήταν να διαβάσει το άρθρο του κανονισμού. Μισό λεπτό. Μια στιγμούλα. Δεν υπάρχει νομικό πρόβλημα. Νομίζω ως προς αυτό συμφωνούμε. Δηλαδή, δυνάμεθα να αναβάλουμε την ψηφοφορία. Είναι αναπόκειται στη διακριτική μας ευχαίρεια. Επί της ουσίας θα αλλάξει τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Θα αλλάξει εντολή. Πιστεύω ότι αν ψηφίσουμε τώρα θα αλλάξει. Γιατί μερικοί έχουν φύγει στο μεταξύ. Οπότε δεν θα έχουμε την ίδια Δεν ε, σωστό να μην έχουμε τη, τον ίδιο σχετισμό δυνάμεων κατά την ψηφοφορία της έκθεσης και μετά κατά την ψηφοφορία της εντολής. Και ο κανονισμός μας καλύπτει. Υπάρχει το δύνατο, όχι το οφείλει να ε, πρέπει να. Οπότε το, θέμα της εντολής ε, εκρεμεί. Και θα το ξαναθέσουμε στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασής μας, ο κύριος Κράμερ. Θα ήθελα να πω ότι ο Γιάκοπ Ταλούντε είπε στην αρχή ότι είναι απαράδεκτο το να λαμβάνει τελευταία στιγμή τον κατάλογο της ψηφοφορίας. Αυτό είναι μικρός παράγοντας, αλλά υπάρχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Η κυρία Τσαπαρδέλ ε, ε, είπε ότι δεν μπόρεσε να γίνει συντονισμός ε, για κάποιες ψηφοφορίες. Καλύτερο θα ήταν να μην γίνουν αυτές οι ψηφοφορίες, ε, να ακολουθήσετε το αίτημα του κυρίου Νταλούντε. Σας παρακαλούμε στο μέλλον να μην κάνετε τέτοιες ψηφοφορίες, διότι όταν λαμβάνουμε τον κατάλογο της ψηφοφορίας τελευταία στιγμή δεν μπορούμε πια να συζητήσουμε το θέμα. Και θα έπρεπε να συμμετέχουν και όλες ε, οι ε, πολιτικές ομάδες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, να το αποτέλεσμα. Κύριε Κράμερ, άκουσε και τον κύριο Νταλούντε, άκουσε και την απάντηση της εισηγήτριας και κανένας στην αίθουσα δεν ζήτησε αναβολή της ψηφοφορίας. Οπότε θα πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί στις βάσεις μας. Εύλογη ήταν η παρατήρηση του κ. Νταλούντε, άκουσα την απάντηση της εισηγήτριας, αλλά κανένας δεν ζήτησε αναβολή της ψηφοφορίας. Και αυτό το αίτημα θα έπρεπε να το θέσουμε σε ψηφοφορία. Ε, και παρόλο που υπήρχε κάποια δυσκολία, τελικά έγινε σεβαστή διαδικασία. Ο κύριος Βαντάλεν. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να μάθουμε από όλα αυτά. Όταν η συγγήτρια πρότεινε μη ψηφοφορία της εντολής, αυτή η πρόταση θα έπρεπε να τεθεί σε ψηφοφορία, αλλά αυτό δεν συνέβη. Άκουσα τις εξηγήσει σας και συμφωνώ ότι έχουμε διάφορες υποχρεώσεις εδώ, πρέπει να κάνουμε τη διάκριση και να επανέλθουμε στο θέμα αργότερα. Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι όταν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, όντως ήταν κάπως ιδιάζουσα ε, κατάσταση στην ψηφοφορία γιατί μερικοί έρχονται μόνο για να ψηφίσουν. Αλλά όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, γιατί να μην προβλέπουμε μια περίοδο προβληματισμού. Καλό κάνει, κακό δεν κάνει. Και δεν πρόκειται να αλλάξει η πολιτική φύση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Απλώς αφήνουμε λίγο χρόνο για να κατασταλάξουμε και να δούμε Άλλωστε όλοι συμφώνησαν να γίνει ψηφοφορία. Η ψηφοφορία έγινε υπό κανονικέ συνθήκες. Η συγγήτρια απεφάνθη προς την εντολή, οπότε θα αφήσουμε λίγο χρόνο για να κατασταλάξουμε, να προβληματιστούμε. Και είπα και στην κυρία Φώστερα, από τη στιγμή που έχει, αλλά, έχει μείνει άδεια μισή αίθουσα, δεν είναι σκόπιμο να γίνει ψηφοφορία για την εντόλη. Και θα αποφύγουμε και περιττές αντιρρήσεις ε, μετά. Περνάμε στο επόμενο λοιπόν σημείο της ημερήσης διάταξης μετά την ολοκλήρωση των ψηφοφοριών. Έκθεση Αγιούτο για συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια για πέντε λεπτά, στην κυρία Ντανιέλα Αγιούτο, για να μας παρουσιάσει τις αδρές γραμμές της εκθεσής της και τις πολιτικές της θέσεις. Κυρία Αγιούτο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ίσως να περιμένουμε λίγο να βγουν όλοι από την αίθουσα. Λοιπόν, εγώ προχωρώ τις εργασίες για τη σχετική οδηγία για τις συνδυασμένε μεταφορές, ε, κάνω και διάφορες συναντήσεις για να λάβω υπόψη όλες τις θέσεις, οι οποίες είναι και από τον κλάδο, αλλά και ε, να λάβω υπόψη και τις εθνικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις των πολιτών ολοκλήρωσα το κείμενο του πρώτου σχεδίου έκθεσης, το οποίο μαζί και με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στόχο έχει να διευκρινίσει καλύτερα κάποιες πτυχές και να περιοτείνει περαιτέρω μέτρα για να υποστηρίξουμε τις συνδυασμένες μεταφορές στην Ευρώπη. Το πρώτο σημείο αφορά ακριβώς τον ορισμό. Θέλησα να κάνω καλύτερη διάκριση μεταξύ οχημάτων ε, με ε, οδηγό και αυτοκινούμενων οχημάτων. Επίσης, για να υπάρχει στο πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας και ε, ε, δυνατότητα για ημι φορτηγά 44 τόνων, ε, προσπάθησα να δώσω κάποιες διευκρινήσει. Όσον αφορά τις οδικές μεταφορές, για να διατηρήσει κανείς τις οριακέ αποστάσεις των 150 χιλιόμετρων σε ευθεία γραμμή, ή ε, το 20% της απόστασης ευθεία γραμμή της συνολικής διαδρομής, προσπάθησα να λάβω υπόψη μου τις ε, πιο κοντινές ή τις πιο κατάλληλες ε, δυνατότητες συνδυασμού. Και επίσης ε, λαμβάνουμε υπόψη μας και τις συνδυασμένες μεταφορές που ξεκινούν εκτός Ευρωπαϊκής, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την περίπτωση, μόνο όταν οι αποστάσεις ε, που καλύπτονται σε αυτή την περίπτωση εντός Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπίπτουν στο πεδίο της εφαρμογής της οδηγίας. Όσον αφορά τα μέτρα για να δώσουμε κίνητρα για συνδυασμένες μεταφορές, έχουμε τη δυνατότητα για διάφορες λύσεις, καταρχάς στήριξη των επενδύσεων. Υπάρχουν επίσης φορολογικές ελαφρύνσεις και κάποιες εξαιρέσεις για τους κλάδους. Οι επενδύσεις είναι απαραίτητες ε, διότι δεν υπάρχει ίση κατανομή σε όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια των διαφόρων υποδομών. Ε, πέραν της αύξησης των τερματικών σταθμών θα πρέπει να βελτιώσουμε και την πρόσβαση στους δερματικούς σταθμούς. Λαμβάνω υπόψη μου βεβαίως και δεν μπορώ, ότι δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά περιμένουμε και από τα κράτη-μέλη να υπάρχει μια δέσμευση και να εγκριθούν κάποια μέτρα για την υποστήριξη των υποδομών, ιδίω αν λάβουμε υπόψη μας ότι με την αναθεώρηση της οδηγίας για την Ευρωβινιέτα θα αυξηθούν ε, τα έσοδα ε, στον κρατικό κορβανά, ακριβώ για να βελτιώσουμε τις ε, ε, βιώσιμες συνδυασμένες μεταφορές. Ως περαιτέρω μορφή στήριξης ε, θα ε, θέλαμε ίσως να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο για κάποιες διευκολύνσεις για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως στις περιπτώσεις που οι επενδύσεις δεν υπερβαίνουν το 35% της συνολικής επένδυσης. Κάποιες άλλες ελαφρύνσεις θα μπορούσαν να προκύψουν από την εφαρμογή μειωμένων τελών για μέσα τα οποία χρησιμοποιούν συνδυασμένες μεταφορές και χρησιμοποιούν και διάφορες τύπους υποδομών. Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι φλέγον ζήτημα είναι το θέμα του καμποτάζ και της απόσπασης των εργαζομένων. Το καμποτάζ είναι ένα μέτρο το οποίο σίγουρα δίνει κίνητρα για συνδυασμένε μεταφορές, αλλά θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια στον ορισμό, ώστε να μην υπάρχουν ε, καταχρήσεις των κανόνων για να, να, για να μπορέσουν να έχουν ε, παράνομο καμποτάζ. Όσον αφορά την απόσπαση των εργαζομένων, Ήμουν σίγουρα υπέρ της εφαρμογής μέτρων για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων των οδηγών για το τμήμα της οδικής μεταφοράς. Τέλος, το θέμα της ψηφιοποίησης. Ελπίζω σύντομα να καταλήξουμε σε μια κατάσταση στην οποία δεν θα χρησιμοποιούνται έγγραφα ε, για να μπορέσουμε να έχουμε πιο γρήγορες διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης. Για τον λόγο αυτό, οι χώρες μελή πρέπει να δέχονται τα έγγραφα όταν ε, παρουσιάζονται σε ηλεκτρονική μορφή. Ο τελικός στόχος είναι να υπάρχει μία ε, συνολική πρόταση με όλες τις πιθανές απαιτήσεις που μπορεί να προκύψει, με προστασία των δικαιωμάτων όλων, αλλά ταυτόχρονα με στόχο να δώσουμε πραγματικά κίνητρα στον τομέα και να υπάρξει ανάπτυξή του. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Θα ακούσουμε τώρα τους και οδησηγητές ε, για το ΕΛΚΣ. και οδησηγητή είναι η κυρία Σμίτ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ε, αρκετά ισορροπημένη προσέγγιση, αν και θα υποβάλουμε τροπολογίες για κάποια θέματα. Επί της αρχής ε, μιλάμε για σχετικά μεγάλο πρόβλημα και για έναν πολύ καλό σκοπό. Είναι φιλόδοξο το σχέδιο διότι οι συνδυασμένες μεταφορές ε, είναι πολύ πιο ε, δαπανηρές και δύσκολες ε, από ότι οι οδικές μεταφορές. Με την οδηγία περί συνδυασμένων μεταφορών διαπιστώνουμε ότι οι συνδυασμένες μεταφορές θα είναι κατά 150% πιο ακριβές από τις οδικές μεταφορές και επίσης ε, έχουμε σημεία συμφόρησης στους τερματικούς ε, σταθμούς μεταφόρτωσης. Χρειάζονται τερματικοί σταθμοί και δρόμοι προσέγγισης ε, και αναφέρομαι στο τούνελ του Μπρένερ καθώς είμαι Αυστριακή. Καταλαβαίνετε ότι χρειαζόμαστε μια ισορροπημένη προσέγγιση, διότι τελικά έχουμε ένα πρόβλημα ε, λοιπούς ε, υποδομής και υψηλότερης τιμής. Εάν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας, ε, θα πρέπει να κάνουμε μαζικές ε, επεμβάσεις ε, στην αγορά και τότε θα ξεκινήσουν τα προβλήματα. Στις οδικές μεταφορές ήδη έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό με τις σιδηροδρομικές μεταφορές, με το άνοιγμα των σιδηροδρομικών μεταφορών πριν από 10 χρόνια είναι ακόμα σχετικά περιορισμένος ο ανταγωνισμός. υπήρχε και ένα πρόβλημα με τη Γαλλία ε, επειδή είχαμε πολύ λίγους ε, οδηγούς συνδρομικών μηχανών ε, που να μιλούν γαλλικά, οπότε δεν μπόρεσαν να παραταθούν, να επεκταθούν οι μεταφορές μέχρι τη Γαλλία. Θα πρέπει να προσέξουμε να φέρουμε τις σιδερόμους στο επίπεδο των δρόμων. Συχνά αναφέρεται ως παράδειγμα η Αμερική. Εκεί λειτουργούν καλά οι συνδυασμένε μεταφορές επειδή λειτουργούν καλά και οι εμπορευματικές μεταφορές. Ως ΕΛΚ στηρίζουμε όλα τα μέτρα που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα των σιδηροδρόμων το να ε, μεταφέρουμε ε, τις μεταφορές ε, στους σιδηρόμους μόνο και μόνο επειδή κάνουμε πιο ακριβές τις οδικές μεταφορές, αυτό δεν αποτελεί σωστή προσέγγιση. Γενικά πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση η έκθεση, αλλά νομίζω ότι η μεταφορά των μεταφορών από τον δρόμο στους σιδηροδρόμους θα είναι δύσκολο να γίνει με ε, την οδηγία αυτή, διότι ε, θα είναι πιο ακριβές οι μεταφορές για τους ε, καταναλωτές και πιο πολύπλοκες για τους εμπόρους. Δεν έχουμε στοιχεία για τις συνδυασμένες μεταφορές. Η ψηφιοποίηση θα πρέπει να προχωρήσει, όπως είπε και η συγγήτρια. Και θα πρέπει να έχουμε εναρμονισμένη εφαρμογή σε όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει να κάνουμε πιο ελκυστικέ τις συνδυασμένε μεταφορές. Υπάρχουν όμως ε, πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμη και στηρίζουμε την πρόταση της εισηγητίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σμιτ. Για του Σοσιαλιστέ και δημοκράτες η κυρία Δελμόντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ε, να ευχαριστήσω Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τη συναδελφό Ντανιέλα Γιούτο για τη δουλειά τη σε έναν τόσο σημαντικό τομέα όπω είναι αυτό των συνδυασμένων μεταφορών. Θέλουμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και να δώσουμε μια περαιτέρω όθηση προς μεταφορές οι οποίε πραγματικά να είναι συνδυασμένε ε, και να χρησιμοποιούν διάφορα μέσα μεταφορά για να μειώσουμε τις οδικές μεταφορές και να είναι πιο αποτελεσματικές ε, όχι μόνο για αποσυμφόρηση της κίνησης αλλά και για μείωση των εκπομπών. Η χορύπανση δε είναι πάρα πολύ σημαντική και τέλος υπάρχει και το θέμα των ατυχημάτων. Θα πρέπει λοιπόν ε, να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογής και στις εθνικές μεταφορές. Αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση σίγουρα της ε, χρήσης των συνδυασμένων μεταφορών και θα υπάρχει και αύξηση και γι' αυτό το σκοπό ε, και γι' αυτό κατά την άποψή μας πρέπει να αλλάξει και ο τίτλος της οδηγίας και πρέπει να διευκρινίζουμε ότι θα πρέπει να γίνεται χρήση των συνδυασμένων μεταφορών και εντός των κρατών μελών για να ε, αυξηθούν οι συνδυασμένες μεταφορές ε, και να μην στοχεύουμε μόνο σε μεταφορές οι οποίες στοχεύουν στις τρίτες χώρες. Εγώ διαφωνώ με το όριο των 150 χιλιόμετρων ή του 20% της απόστασης, γιατί κατά την άποψή μου αυτό είναι ένας τρόπος να δημιουργήσουμε και διαφορετικές ερμηνείες και αυτό δεν θα έπρεπε να δημιουργήσει ακριβώ σύγχυση, ε, δεδομένου ότι ε, μας ενδιαφέρει βελτίωση και να μην υπάρχουν μόνο δικές μεταφορές. Θα έπρεπε ίσως να υπάρχει ένα πιο σαφές κριτήριο, για παράδειγμα καθορίζοντας αυτό το όριο στα 200 χιλιόμετρα, αλλά να θεωρούνται ε, πραγματικά τα 200 χιλιόμετρα της οδικής απόστασης. Επίσης είμαι υπέρ της περαιτέρω για τη διαβίβαση των ε, ε, εγγράφων των συνδυασμένων μεταφορών, τα οποία θα πρέπει να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά. Όσον αφορά τα οικονομικά κίνητρα, πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις πραγματικές απαιτήσει των κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Τελμόντε. κύριος Ζωτόφσκι για το ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα εκ μέρους της ομάδας ECR να <clears throat> ευχαριστήσω την κυρία Γιώτο για την ε, εκπόνηση της έκθεσης. Γιατί δίνει μια πολύ καλή απάντηση στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταρχήν. Συμφωνούμε απόλυτα με την πρόταση ότι οι συνδυασμένε μεταφορές θα πρέπει να αναπτύσσεται χάρη στην επικέντρωση της προσοχής μας σε τρία θέματα. Προσδιορισμό των ορισμών των όρων και των εξαιρέσεων, κατάλληλων επενδύσεων στις υποδομές και την ψηφιοποίηση της διαδικασίας του ελέγχου. Βέβαια, υπερβολικά φιλόδοξες προτάσεις στα θέματα τα κοινωνικά ίσως δημιουργήσουν φραγμό στην ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών. Ε, ε, για τις οποίες το δικό τμήμα εξακολουθεί να έχει μεγάλη σημασία. Και κυρίως ε, είμαστε κατά της υπερβολικής γραφειοκρατίας που δημιουργεί ε, επιβαρύνσεις στους επιχειρηματίες και αύξηση του κόστους και σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με την ελεύθερη διακίνηση των υπηρεσιών. Ε, κατά τη δική μας ε, άποψη, η συμπερίληψη των οδικών μεταφορών στις συνδυασμένες μεταφορές, ε, ιδιαίτερα για τους αποσπασμένους ε, αποσπασμένους με βάση την οδηγία 96 του 94 δεν είναι αποδεκτό. Και ελπίζω στα πλαίσια το συζητήσω και των διαπραγματεύσεων με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες να καταλήξουμε σε λιγότερο περιοριστικές διατάξεις και πιο φιλικές προς τις επιχειρήσεις των μεταφορών. Σας ευχαριστούμε κυρία Ζωτόφσκη. Η ε, κυρία Μπιλμπάο για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε, καλημέρα συνάδελφοι. Καταρχήν ε, συμφωνούμε και εμείς ε, και ευχαριστούμε την εισηγήτρια για τις προσπάθειές της και συμφωνούμε ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τους ορισμούς και τις πιθανές εξαιρέσεις Και όπως είπαμε και στην πρώτη παρέμβαση, ε, κάθε χώρα διαφορετικά ερμηνεύει τις συνδυασμένες μεταφορές, οπότε θα πρέπει πρώτα να συμφωνήσουμε ως προς τον ορισμό. Τι εστί συνδυασμένη μεταφορά. Συμφωνούμε ως προς την ανάγκη ενίσχυσης της ψηφιοποίησης του συστήματος, χρησιμοποιώντας ε, την τεχνολογία και τα ηλεκτρονικά μέσα για να ε, ελαφρύνουμε το γραφειοκρατικό άχθος και τις διατυπώσεις και να διευκολύνουμε τις συνδυασμένες μεταφορές. Συμφωνούμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση και στις επενδύσεις, αλλά ταυτόχρονα συμφωνούμε ότι θέλουμε και άλλες πληροφορίες ως προς την ύπαρξη των υποδομών, γιατί κάποιοι από τον κλάδο, τουλάχιστον σε κάποιες χώρες, μας λένε ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις, που προσπαθούμε επίσης να ευνοήσουμε και να παροτρύνουμε ε, ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, αναχαιτίζονται όταν παράλληλα γίνονται και δημόσιες επενδύσεις. Δηλαδή, καλό θα ήταν να μην εκτελούμε νέες επενδύσεις όταν δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς οι υπάρχουσες υποδομές. Σε ό,τι φορά τις ενδομεταφορέ, ε, το καμποτάζ δηλαδή και τους αποσπασμένους ε, οδηγού ε, ή τους μετακινουμένους, θα πρέπει να δούμε παράλληλα το θέμα των οδικών μεταφορών και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε εκεί στο θέμα του καμποτάζ, τον ορισμό του καμποτάζ και τους αποσπασμένους εργαζόμενους δεν μπορούμε να απομονώνουμε τις εκθέσεις, θα πρέπει να τις εξετάσουμε εκ παραλλήλου και να συμπεριλάβουμε στην έκθεση αυτή την πρόοδο που γίνεται στα θέματα του καμποτάζ των Εδωμεταφορών. Επίσης, συμφωνώ ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μας δώσουν πιο ακριβείς και λεπτομερικές πληροφορίες, γιατί μας λείπουν στοιχεία και στατιστικά δεδομένα για να ε, δημιουργήσουμε σαφή εικόνα για τον κλάδο, για την πρόοδο των τελευταίων χρόνων και επίσης ε, για την ενίσχυση του ελέγχου. Σε ό,τι αφορά τα κίνητρα, τα ενάβσματα για τη χρήση των συνδυασμένων μεταφορών. Και σε αυτό το θέμα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρώτα θα πρέπει να ορίσουμε τα υπόλοιπα ζητήματα. Και επαναλαμβάνω την ανάγκη να έχουμε συνεπτικές συνδυασμένες μεταφορές με τα μέτρα που έχουμε ήδη ε, υιοθετήσει και τα στρατηγικά σχέδια που έχουν εφαρμόσει τα κράτη-μέλη. Είμαστε υπέρ της συνοχής και κατά την εκτέλεση ε, και την τήρηση των προθεσμιών, με τα TNT για παράδειγμα, τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Γιατί σε μερικές χώρες τα διευρωπαϊκά δίκτυα των μεταφορών προχωρούν με καλούς ρυθμούς και πιστεύω ότι οι συνδυασμένε μεταφορέ δεν θα λειτουργήσουν εύρυθμα και δεν θα αναπτυχθούν ε, επαρκώ αν δεν απαιτήσουμε και πάλι από τα κράτη-μέλη μια συνοχή σε όλες τις πτυχές των μεταφορών. Υπό το πνεύμα αυτό έχω καταθέσει και κάποιες τροπολογίες για να βελτιώσουμε σε συνεργασία με τους άλλους συναδέλφους την έκθεση. Και φαντάζομαι θα επαναλάβουμε την μέχρι τώρα καλή προσπάθεια της κυρίας Αγιούτο. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπιλμπάου. Ο κύριος Νταλούντε από τους Πράσινους. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Αγιούτο για το σχέδιο έκθεσης που ήδη περιέχει πολλά θετικά στοιχεία. Θα θέλαμε όμως περαιτέρω ε, αποσαφήνιση της φιλοδοξίας, της αύξησης των μέγιστων ορίων, καθώς και τη δυνατότητα εκ των υστέρων ελέγχων. Επίσης ε, δεν ε, συμφωνούμε με την ε, εξαίρεση των οδικών μεταφορών από τους κανόνες περί ενδομεταφορών, διότι αυτό υπονομεύει τους κανόνες αυτούς. Είναι πολύ σημαντικό να ξεφύγουμε από τις οδικές μεταφορές. Θα θέλαμε καλύτερη ενσωμάτωση των εσωτερικών πλωτών οδών και γενικότερα της ναυσιπλοείας, στο, της στο κείμενο του, της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Madame Κυρία γκραντς ζήτησε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήδη ε, είπαμε ότι ο στόχος ε, είναι να έχουμε πιο περιβαλλοντικές μεταφορές, δηλαδή να ξεφύγουμε από τις οδικές μεταφορές. Ε, δεν είναι πολύ απλό το θέμα αυτό. Αντιθέτως, ε, προβλέπεται εδώ πέρα σημαντική απελευθέρωση των μεταφορών και έτσι θα γίνουν πιο ελκυστικές οι οδικές μεταφορές ε, και δεν το θέλουμε αυτό. Θα υποβάλουμε σχετικές ε, τροπολογίες. Έχουμε ήδη αναφέρει το 20% της ολικής διαδρομής καθώς και την ακτίνα που περιγράφεται εδώ πέρα για τις μεταφορές. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των εργαζομένων και στη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα είχαμε σχετικές συζητήσεις. Η απόσπαση και οι ενδομεταφορές είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε και θα πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρχουν εξαιρέσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Αν δεν θέλει άλλος κανείς το λόγο, θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση ΜΟΥΒ. Ο κύριος Ανταπέντο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σχολιάσω την έκθεση που χαιρετίζουμε ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η στριπτική πλειοψηφία των τροπολογιών της ηγητρίας ε, στόχο έχουν τη διευκρίνηση ή την ενίσχυση των διατάξεων ε, της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, με βάση τους στόχους της περαιτέρω προώθησης της χρήσης των συνδυασμένων μεταφορών, της παρότρησης των κρατών μελών να ενισχύσουν τη στήριξη προς τις συνδυασμένες μεταφορές και να πλουστεύσουν τους κανόνες, να ενισχύσουν την εφαρμογή των κανόνων και να αποτρέψουν τις καταχρήσεις. Αυτή είναι η στόχη μας. Οπότε με αυτό το πνεύμα χαιρετίζουμε ιδιαίτερος τις τροπολογίες που διατηρούν τον ορισμό και προβλέπουν και τη δυνατότητα της ε, διαφύλαξης της πρόσβασης στον ε, κοντινότερο ε, σιδηροδρομικό σταθμό αν δεν υπάρχει άλλο σταθμό στα πλαίσια των, στο, στην ακτίνα των 150 χιλιόμετρων. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα της ακτίνας γιατί μια αυστηρή, αυστηρή χρήστη ε, της χρήσης των οδικών μεταφορών ίσω έχει τον επιθύμητο αποτέλεσμα τη μεταφορά και πάλι των φορτηγών στις αυτοκινητοδρόμου αντί να δίνει κίνητρα για τι ιδιασμένες μεταφορέ. Επίση, χαιρόμαστε για την ενίσχυση τη διάταξη περί ψηφιοποίηση, γιατί θεωρούμε ότι η ψηφιοποίηση θα βοηθήσει ιδιαίτερω για την αποφυγή των καταχρήσεων ώστε όντως η επιχείρηση να είναι συνδυασμένη η επιχείρηση μεταφοράς και να μην χρησιμοποιείται το, ως παραθυράκι, ως πρόσχημα. Και επίσης ε, συμφωνούμε με την πρόταση για περαιτέρω υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων από τα κράτη-μέλη και τουλάχιστον ένα μέτρο τέτοιο να είναι υποχρεωτικό μέτρο στήριξης. Έτσι θα παρατρύνουμε τα κράτη-μέλη να ε, υποστηρίξουν πιο ενεργά τις συνδυασμένες μεταφορές. Ένα θέμα των τροπολογιών που δεν, δεν αναφέρθηκε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κοινοποίηση των ε, κρατικών ενισχύσεων ή το θέμα της απόσπασης των εργαζομένων, τα σημειώνουμε. Σε ό,τι αφορά τους κοινωνικούς κανόνες, φυσικά ισχύουν και για τις συνδυασμένες μεταφορές γιατί κρίνουμε σκόπιμο και σημαντικό να κρατήσουμε μια συμμετρία μεταξύ των κανόνων που ισχύουν για τις διεθνείς ιδιασμένες μεταφορές και αυτών που ισχύουν για τις ε, διεθνείς οδικές μόνο μεταφορές. Γιατί αυτές είναι οι δύο διαφορετικές δραστηριότητες ε, που είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους, οι διεθνείς συνδυασμένες και οι διεθνείς αμυγός οδικές μεταφορές. Ευχαριστώ για τις προτάσεις. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τώρα η συγκεκριά μας και πάλι η κυρία Αγιούτο για τα συμπεράσματα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα όσα είπαν όσον αφορά τα όσα έκανα μέχρι τώρα και θα ήθελα μισό λεπτό να σταθώ λίγο σε κάποιες παρατηρήσεις που έγιναν. Όσον αφορά την όλη συζήτηση για τους εκτονιστέρων των ελέγχους, οι εκτονιστέρων έλεγχοι δεν έρχονται να προσθεθούν και χάθηκε το μικρόφωνο της ομιλήτριας. Δεν ακούσατε τίποτα, φαντάζομαι, να τα ξαναπώ από την αρχή. Λοιπόν, όσον αφορά την όλη συζήτηση των εκτονιστέρων ελέγχων, δεν πρόκειται για προσθήκη. Απλώς ε, αντιλαμβανόμαστε ότι κάποια έγγραφα πολύ εύκολα μπορεί να δοθούν μετά από την ε, μεταφορά, για πρακτικούς λόγους και έτσι απλώς θέλουμε να διευκολύνουμε λίγο το γραφειοκρατικό άχθος, το οποίο ε, είναι τμήμα των κινήτρων που θέλουμε να παρέχουμε σε αυτή την περίπτωση. Όσον αφορά τους φόβους ε, ότι μπορεί να δώσουμε ουσιαστικά ένα ελευθέρας ε, και πλήρη απολευθέρωση των ε, οδικών μεταφορών, είναι ακριβώς το αντίθετο αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Εμείς προσπαθούμε όσο το δυνατόν τα εμπορεύματα να γίνονται μέσω σιδηροδρόμων και ακριβώς λόγω σχεδιασμού περιμένουμε ότι θα υπάρξει αυτή η μετάβαση επιτρέψαμε ουσιαστικά να μεταφέρονται ε, μέσω οδικών δικτύων το τελευταίο τμήμα της μεταφορών και ακριβώς ε, ο στόχος είναι να δώσουμε κίνητρα και να πιέσουμε να επιλέγεται αυτή η οδός. Να υπενθυμίσω ότι αν δεν δώσουμε κίνητρα για τις συνδυασμένε μεταφορών, ε, μεταφορές, σήμερα τα εμπορεύματα μεταφέρονται αποκλειστικά και μόνο μέσω οδικών δικτύων γιατί είναι πολύ πιο βολικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί φόβοι βεβαίω, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε οι επιχειρήσεις να επιλέγουν ε, και άλλα μέσα μεταφοράς. Κατά τα λοιπά, περιμένω να διαβάσω τις τροπολογίες σας και φυσικά ε, θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε ώστε να προτείνουμε ένα κείμενο το οποίο θα είναι όσο το δυνατόν πιο πλούσιο ώστε αυτές οι συνδυασμένες μεταφορών, μεταφορές να λάβουν και την όφηση που τους αξίζει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γιούτο. Με αυτό ολοκληρώνω τη συζήτηση. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 16 Μαΐου 2018. Ώρα δεν έχει εδώ, ε. Στις 12. 16 Μαΐου λοιπόν 2018, 12 η ώρα, ψηφοφορία στην Επιτροπή στις 10 Ιουλίου. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Η έκθεση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών αναδιατύπωση του προηγούμενου κανονισμού, να δώσω αμέσως το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Λιμπεράτσκι, τον οποίο τον είδα εδώ να περνάει. Α, Ωραία. Μπόγκουσλαβ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Ντομινίκ. Θα είμαι λακωνικός. Καταρχήν, έχετε αυτό το έγγραφο, μόνο 190 σελίδες. Ε, και περιλαμβάνει 600 περίπου τροπολογίες. Οι βασικοί τομείς που εντοπίστηκαν αναλύθηκαν στις ζητήσεις με σκιώδη ηγητές, ε, ενδιαφερόμενους. Είχαμε περίπου 20 διαφορετικές ε, συνεδριάσεις, γεύματα εργασίας, συζητήσεις με ενδιαφερομένους και με σκιώδεις ηγετές. Καταρχήν, ε, υπάρχει μεγάλη προβολή του συγκεκριμένου κανονισμού. Συμφωνούμε ότι μιλάμε για δισεκατομμύρια ανθρώπους που επηρεάζονται άμεσα κάθε χρόνο από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Δεύτερο, θέλουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση, δηλαδή θα πρέπει να εγγυηθούμε την ποιότητα των υπηρεσιών να θεσπίσουμε κάποιες υποχρεώσεις για τους παρόχους υπηρεσιών, αλλά ταυτόχρονα να διαφυλάξουμε την ικανότητα της παροχής των υπηρεσιών. Δηλαδή, θέλουμε κάποια μέτρα, κάποιες διατάξεις και κανονισμούς, ρυθμίσεις που θα επιτρέπουν στις σιδηροδρομικές ε, επιχειρήσεις μεταφορών να ε, δρούν αποτελεσματικά και να προστατεύσουμε και τους επιβάτες. Γιατί αυτό ζητούν οι συμπολίτε. Και πρόθεσή μα είναι να προστατεύσουμε του επιβάτε, να προστατεύσουμε του πολίτε, αλλά ταυτόχρονα πρόθεσή μα είναι να μην βλάψουμε, να μην πλήξουμε του παρόχου υπηρεσιών, του μεταφορεί. Εδώ έχουμε τρία μέρη. Αυτού που μεταφέρουν τους επιβάτες, αυτούς που ε, προσφέρουν υπηρεσίες στα πλαίσια των υποδομών, ιδιαίτερα σιδηροδρομικούς σταθμούς και εκείνους που πολλούν εισιτήρια. Ε, επίσης, ε, λαμβάνουμε υπόψη τα συμφέροντα των ατόμων με αναπηρία μειωμένη κινητικότητα. Πολύ σημαντικά θέματα αναφέρονται στο συγκεκριμένο κανονισμό και για την προάσπιση των δικών τους δικαιωμάτων. Είμαι ευγνώμων προς τους ε, σκιώδεις ηγητές και τους συμφέροντοχους για τη συνεργασία που είχαμε, αλλά και την ε, συνεργασία που είχαμε με μονομένους ε, ευρωβουλευτές που είναι μέλη της Επιτροπής μας και που συνέβαλαν στη διαμόρφωση έκθεσης. Εγώ προσβλέπω σε μια αγαστή και αποτελεσματική συνεργασία κατά τη διαμόρφωση αυτής της έκθεσης και την εκπόνηση συμβαστικών τροπολογιών. Πάντως, η δική μου ιδέα είναι να έχουμε μια ισορροπημένη πρόταση για έναν ισορροπημένο καλό, άρτιο κανονισμό που θα αυξήσει το μερίδιο των σιδηροδρόμων στην αγορά των μεταφορών. Δηλαδή θα προσελκύσουμε επιβάτες στους σιδηροδρόμους, σιδηροδρομικές μεταφορές και θα επιτρέψουμε στους, στις υπηρεσίες ε, σιδηροδρομικών μεταφορών να παρέχουν, ε, στις επιχειρήσεις σιδηροδρομικών μεταφορών να παρέχουν πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες. Ευχαριστώ Μπογκουσόφ. Θα ακούσουμε τώρα τους και οδησηγητές των διαφορών ομάδων. Δόκτωρ Μιζελία πρώτα από το ΕΛΚ. Ε, Ρενό, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ ε, για την ε, εισαγωγή και την αναφορά του τίτλου μου. Ε, όντως έχω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ιατρικό για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την εισαγωγή. Πάνω από 600 τροπολογίες κατατέθηκαν πολύ περισσότερες δηλαδή από το σύνολο του, της δέσμης ε, κινητικότητας. Σίγουρα ε, οι επιβάτες μας έχουν πληγεί από τις ε, ε διαδοχικές απεργίες ε, των σιδηροδρόμων. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε προστασία του κλάδου αυτού και των επιβατών. Είναι ελπιδοφόρες οι τροπολογίες και σίγουρα θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον εισηγητή για να καταλήξουμε σε, σε συμβαστικές πρωτοβουλίες ώστε να ληφθούν υπόψη οι φιλοδοξίες και οι προσδοκίες των επιβατών μας. Τα, πιο, τα τέσσερα πιο σημαντικά σημεία του κανονισμού καλύφθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις τροπολογίες ε, χαίρομαι για τη φιλοδοξία που έχουν επιδείξει κάποιε τροπολογίε, ιδιαίτερα στην πρόταση να ενισχυθεί αισθητά η προσβασιμότητα στο σιδηροδρομικό δίκτυο των ε, ατόμων με αναπηρία και η μειωμένη κινητικότητα. Μια σύντομη επισκόπηση. Η πρωτοχική στόχη των τροπολογιών είναι πρώτον, ε, η εφαρμογή του συνόλου του κανονισμού και χωρί εξαιρέσει από το 2019. Πολλές τροπολογίες ζητούν διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή ώστε να καλύψει και τις περιφερειακές σιδηροδρομικές υπηρεσίες. Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί αυτό ζητώ από την αρχή των εργασιών. Και το να αφήσουμε περίπου 90% των επιβατών στη μοίρα τους είναι απαράδεκτο και χαίρομαι για την πρόταση αυτή, για την επέκταση του περίοδου εφαρμογή. Δεύτερον, βελτιώνουμε την προσβασιμότητα των 80 εκατομμυρίων ε, συμπολιτών μα που έχουν μειωμένη κινητικότητα ή αναπηρία ό,τι φορά του σιδηροδρόμου. Και αυτό είναι ε, κοινό στόχο όλων των πολιτικών ομάδων. Επίση, προκοινοποίηση. Ε, για συγκεκριμένες ώρες. Αυτό ήδη γίνεται στο Βέλγιο και στη Δανία για να διευκολυνθεί η καθημερινότητα των συμπολιτών μας που έχουν κατεξοχή ανάγκη από τέτοιες δημόσιες ε, συγκοινωνίες και μεταφορές. Επίσης, θα πρέπει η κοινοποίηση να σχετίζεται με την ε, συχνότητα συγκεκριμένων διαδρομών. Πάντως, ε, στα πλαίσια των συμβαστικών τροπολογιών θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και από τους διαχειριστές του σιδηροδρόμου και από τους επιχειρηματίες μεταφορών να προβλέψουν πιο φιλόδοξες, διατά... πιο φιλόδοξες ρυθμίσεις. Επίσης, το θέμα της αποζημίωσης ε, για ματέωση ή καθυστέρηση. Ε, μειώνεται το κατόφλι στα 30 λεπτά. Ε, σε κάθε περίπτωση πάντως ε, συμφωνούμε ως προς τη διάγνωση. Μία ώρα καθυστέρηση για αποζημίωση 25% του εισιτηρίου για μία διαδρομή διορών είναι υπερβολικό. Ενώ αν μειώσουμε στα 30 λεπτά θα, ε, τον, ε, την ώρα καθυστέρηση για το δικαίωμα αποζημίωση είναι ένα μήνυμα προ επιβάτε και τι επιχειρήσει Για να σταματήσει αυτή η πολιτική των αλλεπάλληλων καθυστερήσεων. Τέταρτος στόχο. Ενιαίο εισιτήριο. Έχει κεντρική θέση στι συζητήσει. Θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να βρούμε συμβαστική λύση μεταξύ εκείνων που ζητά υποχρεωτικό στι πωλήσει ενιαίου εισιτήριου και εκείνων που δεν θέλουν ούτε κουβέντα για το θέμα αυτό. Να βρούμε τη χρυσή τομή. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των επιβατών στη χρήση των σιδηροδρόμων, ε, αναλαμβάνοντας περισσότερες ευθύνες. Και αν γίνει το ολοκληρωμένο εισιτήριο όλο και πιο αυτοματοποιημένο, δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο βάρος των ε, μεταφορέων. Γι' αυτό καλό θα ήταν να εισάγουμε την αρχή της ε, της υπευθυνότητα. Δηλαδή, ο πολιτής των εισιτηρίων θα πρέπει να εξακριβώσει ότι ανταποκρίσεις είναι λογικές. Αλλιώ θα μπορεί ο επιβάτης να στραφεί και προς τον πολιτή εισιτηρίο και να ζητήσει αποζημίωση. Αυτά εκ μέρου του ΕΛΚ και σίγουρα είναι θέμα αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να λάβουμε υπόψη τις προσδοκίε των επιβατών και να κρατήσουμε μια φιλόδοξη κατεύθυνση για να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των επιβατών ε, στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Και ευχαριστώ και πάλι και συγχαίρω τον εισηγητή για το αξιόλογο έργο του σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Πορέμπα για το ECR. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμότατα τον εισηγητή μας, τον κύριο Λιμπεράτσκι, για την πολύ ισορροπημένη και ορθολογική του προσέγγιση στην έκθεση που αφορά τα προβλήματα και τις προσδοκίες των χρηστών σιδεροδρόμων. Θα πρέπει να αποφύγουμε τις υπερβολικές επίσης επιβαρύνσεις των μεταφορέων σιδηροδρομικών, των επιχειρήσεων σιδηροδρομικών μεταφορών. Έχω κάποια σχόλια και ελπίζω μερικές από τις τροπολογίες μας να καλυφθούν από τις συμβαστικές τροπολογίες που θα προτείνει ο εισηγητής. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι ιδιαίτερος που έγινε δεκτή η προθεσμία του 2024 σε ό,τι αφορά τις διατάξεις του κανονισμού 1371 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει το 2020, κάτι που κατά τη γνώμη είναι τοπικό μη ρεαλιστικό και αποκλείεται να εφαρμοστεί. Συμφωνώ με την προθεσμία του 2024. Επίσης, το θέμα της ανωτέρας βίας. Προσπάθησε να βρει μία ισορροπία ο εισηγητής, όχι μόνο για τα θέματα των θεομηνιών ή φυσικών καταστροφών. Αλλά, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να διευρύνουμε τον ορισμό της ανωτέρας βίας και να καλύψουμε και τις τρομοκρατικές ενέργειες ή ενδεχομένως κάποιες απεργίες ή ε, ατυχήματα που οφείλονται στην ε, δράση τρίτων στις ε, ράγες για παράδειγμα. Και το να περιορίζουμε την ανωτέρα βία μόνο στις θεομηνίες και τις φυσικές καταστροφές είναι πολύ περιοριστικό και στενή ερμηνεία. Σε ό,τι αφορά το ενιαίο εισιτήριο, σίγουρα είμαστε υπέρ και θέλουμε να προωθήσουμε την ιδέα του ενιαίου εισιτηρίου. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει πολύ πιο συγκεκριμένα να περιγράψουμε τον μηχανισμό του ενιαίου εισιτηρίου ή την ανάληψη κοινών δράσεων των επιχειρήσεων μεταφορών. Γιατί δίνουμε την εντύπωση ότι κάποιος που αγοράζει μεμονωμένα το εισιτήριο χωρίς ενημέρωση του, στόχου του ταξιδιού, μπορεί να ε, το σε ενιαίο εισιτήριο και να δικαιολογήσουν την απέτηση αποζημίωσης του επιβάτη. Αυτό θα πρέπει να το συγκεκριμενοποιήσουμε περαιτέρω το πώς λειτουργεί το ενιαίο εισιτήριο, γιατί δεν προσδιορίζεται παρκώς προς το παρόν. Σας ευχαριστώ θερμότατα εκ μέρους και των ατόμων με αναπηρία, γιατί εγκύψατε στο ζήτημα των ατόμων αυτών με μειωμένη κινητικότητα και αναπηρίες, ενισχύοντας την πρόσβασή τους. Έχω μία μόνο παρατήρηση για το θέμα αυτό για να αποφύγουμε την εντύπωση ότι θέλουμε οι σιδηρόδρομοι αμέσως να προσαρμοστούν στις ανάγκες των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και αναπηρία. Θα χρειαστούν και οι επιχειρήσεις μεταφορών κάποιο χρόνο για να ετοιμαστούν και να εφαρμόσουν αυτές τις διατάξεις της ενισχυμένης προσβασιμότητας. Αυτά και ευχαριστώ. Προσβλέπω στη συνέχιση της αγαστής συνεργασίας. Πάντως το ECR είναι γενικώ ικανοποιημένο με την έκθεση. Και ελπίζω να καλύψετε τις ε, προτάσεις που σας έκανα με τις συμβαστικές σας τροπολογίες, κύριε Σιγητά. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πορέμπα. Για τους φιλελεύθερους, ο Ματιέ θα μιλήσει αναπληρώνοντας τον Σκέδη Σιγητή. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Σκιώδης Γιάννης δεν μπορεί να είναι παρόν σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν να μεταφέρω κάποια μηνύματά του. Προσβλέπει στις συμβαστικές τροπολογίες και ελπίζει να αντικαταπτρίζουν τις ανησυχίες της ΑλΔΕ που εκφράστηκαν κατά την τελευταία συνεδρία των σκιωδών εισηγητών. Η ΑλΔΕ πιστεύει πρώτον ότι αν δεν επικεντρωθούμε στους επιβάτες κατά την αναθεώρηση αυτής της νομοθεσίας, δεν θα αξίζει τον κόπο πια να μιλάμε για ε, κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών. Ε, ο εισηγητής, ε, μάλλον ο θα πρέπει να προχωρήσουμε πέρα από αυτό που ε, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα πάνω σε τρία θέματα. Καταρχάς όσον αφορά ε, τα συνδυασμένα εισιτήρια. Θα πρέπει αυτά να γίνουν πραγματικότητα και οι επιβάτες ακόμα και αν έχουν ξεχωριτά εισιτήρια θα πρέπει να θεωρείται ότι ε, είναι ένα ενιαίο εισιτήριο όσον αφορά τα δικαιώματά του. Επίσης θα πρέπει να μετριαστούν, ε, να μειωθούν ε, οι καθυστερήσεις ε, και αυτό θα βοηθήσει και την ελκυστικότητα του συνδρομικού τομέα. Τρίτη παρατήρηση για τις εξαιρέσεις στην εφαρμογή αυτού του κανονισμού. δεν θα πρέπει να ισχύουν πια. Εκ μέρους του Γένς, λοιπόν, υπάρχει δυσκολία κατανόησης διότι είναι δύσκολο να εξηγήσουμε κάποια πράγματα στους ψηφοφόρου μας ε, εφόσον οι συνδρομικές ε, επιχειρήσεις ε, είναι και επιδοτούμενες από τα κράτη. Και ιδιαίτερα για επιβάτες που ταξιδεύουν εκτός του κράτου μέλους τους θα πρέπει να γίνει πιο εύκολη η υποβολή παραπώνων με ειδικό έντυπο. Θα πρέπει οι επιβάτε να μπορούν να χρησιμοποιούν τέτοιο έντυπο αντί για αυτό που παρέχουν ε, οι μέρους ε, συνδρομικές επιχειρήσεις. Και θα πρέπει να έχει την ίδια ισχύ αυτό το κοινό έντυπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Γέννης προσλέπει στη συνέχιση των εργασιών ε, και με τον εισηγητή και με τους σκιώδεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε τώρα το λόγο για τους πρασίνους στον κύριο Κράμερ. Μάικολ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους Κιώδης για την πολύ καλή συνεργασία. Σε πολλά θέματα έχουμε ε, ε, την ίδια θέση, σε κάποια άλλα θέματα υπάρχουν διαφωνίες, αλλά αυτό φυσιολογικό είναι μιλάμε για τα δικαιώματα των επιβατών, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στους επιβάτες και όχι στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Άσχετα από το πόσο υψηλό είναι το κόστος της αποζημίωσης, εάν φεύγει στην ώρα του το τρένο δεν χρειάζεται να πληρώσει κανείς αποζημίωση. Ε, στην Γερμανία όμως η κατάσταση έχει ε, φτάσει σε τέτοια όρια που λένε ότι δεν πειράζει, καλύτερα να χρησιμοποιήσω όλα τα τρένα, να μην έχω κάποιο τρένο ρεζέρβα σε περίπτωση ε, προβλήματος. Ε. Ή επίσης ούτε ανάπτυξη των σταθμών. Τεράστιες δαπάνες και μεγάλες καθυστερήσεις. Θα πρέπει λοιπόν πιο μακροπρόθεσμα να σκεφτούν οι συνδρομικές επιχειρήσεις. Η ανωτέρα βία φυσικά είναι σημαντικό θέμα. Γνωρίζουμε πώς έχουν τα πράγματα στις αεροπορικές μεταφορές. Σε, κάθε, σε κάποιες αεροπορικές επιχειρήσεις σε κάθε καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερα βία. Από τα 26 κράτη-μέλη που έχουν ε, ε, καθυστερήσεις ε, θα έπρεπε να έχουν πληρωθεί 1,5 εκατομμύρια, κάτι που δεν είναι και ψίχουλα. θα μπορούσαμε να λύσουμε το πρόβλημα με μια ασφάλιση που δεν στοιχίζει και πάρα πολλά, ε, ε, έναν εκατό του ειστηρίου. Ε, δεν χρειάζεται λοιπόν να αλλάξουμε τίποτα όσον αφορά την ε, ανωτέρα βία. Όσον αφορά τις, τα ενιαία εισιτήρια, τα through tickets, τις, στα νυχτερινά τρένα έχουν ε, μια ενδιάμεση λύση. εάν δηλαδή χάσει κανείς το τρένο του μπορεί να πάρει το επόμενο. Αυτό ίσχυε, αλλά δεν ισχύει πια. Γιατί, ε, διότι υπάρχει τώρα ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία που λέει ότι για να μιλάμε για through ticket πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο εισιτήριο μπορούμε όμως να πούμε ότι αν η ώρα αναμονής, ε, η ώρα μεταβιβίβασης ε, δεν υπερβαίνει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τότε μιλάμε για ενιαίο εισιτήριο. Ένα από τα αγαπημένα μου ε, θέματα είναι αυτό που έχει κάνει η Αυστρία εδώ και πολύ καιρό, το να ε, παίρνει κανείς μαζί του το ποδήλατο στο τρένο. Γιατί είναι τόσο σημαντικό το θέμα αυτό. Ε, διαπιστώσαμε ότι τα εισιτήρια, ε, ότι τα λεωφορεία έχουν κλέψει το 12% των επιβατών των σιδηροδρόμων επειδή είναι πιο φθηνά. Μόνο γι' αυτό όμως όχι, επειδή μπορούν να πάνε και το ποδήλατο μαζί έχουν χάσει οι σιδηρόδρομοι πάρα πολλούς επιβάτες επειδή ε, δεν ε, επιτρέπουν ε, να πάρουν το ποδήλατο μαζί τους οι επιβάτες. Γιατί χάνετε λοιπόν τους καλύτερους επιβάτες με τον τρόπο αυτό. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να είναι υποχρεωτικό σε όλη την Ευρώπη. Στην Σουηδία ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, σχετικά παράπονα. Ε, βλέπουμε ότι ε, αυξάνονται οι υποδηλάτες, θα πρέπει λοιπόν να τους λάβουμε υπόψη μας. Δεν καταλαβαίνω αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα να πρέπει 24 ώρες πριν να υποβάλουν κοινοποίηση. Θα πρέπει να έχουν ακριβώς τα ίσα δικαιώματα με τους ε, άλλους επιβάτες. Ε, οι Βέλγοι και οι ε, Ολλανδοί απαιτούν ειδοποίηση μία ώρα πριν. Αυτό θα πρέπει να μπορούμε να το κάνουμε σε όλη την Ευρώπη. Σε κάποιε ε, χώρε, ε, εάν ε, κάποιο άτομο με μειωμένη κινητικότητα χρειάζεται σύνοδο, μπορεί να τον πάρει μαζί του δωρεάν, αλλά με το που περνάει τα σύνορα θα πρέπει ξαφνικά να πληρώσει για το άτομο αυτό. Και διάβασα ότι είναι αδύνατες οι διασυνοριακές συνδέσεις στους σιδηροδρόμους για λόγους οικονομίας ε, και φτάνουν τα ε, τρένα στα σύνορα και δεν μπορούν ε, να προχωρήσουν. Πρέπει να σκεφτούμε με ευρωπαϊκό τρόπο τουλάχιστον τα τρένα να μπορούν να πάνε μέχρι τον επόμενο σταθμό. Και επίσης ε, θα πρέπει τα παράπονα να μπορούν να αποστέλλονται ε, από το διαδίκτυο και όχι απαραίτητα στην ίδια τη χώρα, στην επίσημη γλώσσα της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κράμερ. Για την ΚΟΕ η κυρία Γκονζάλης Πένιας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Για την ομάδα μας αυτή η συζήτηση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών είναι ε, θεμελιώδου σημασία. Αν θέλουμε να δούμε τα ποσοστά χρήσης ε, των σιδηροδρόμων για λόγους ε, υγεία, δημόσια ασφάλεια και σεβασμού του περιβάλλοντο να αυξάνονται, πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και κυρίω φιλόδοξοι στα όσα υποσχόμαστε στου χρήστε. Θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε, να έχουμε μια στρατηγική και να προσαρμοστούμε στι σημερινέ ανάγκε και να ε, προετοιμαστούμε και για αυτέ οι οποίε μπορεί να ανακύψουν ε, την επαύριο. Έχουμε υποβάλει τροπολογίε από πλευράς ομάδος ε, για να μεγιστοποιήσουμε, για παράδειγμα, τις διαθέσιμε πληροφορίες σε ανα πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι χρήσει ε, ε, των χρηστών με, και τη δυνατότητα να έχουν και το ποδήλατό τους, να δώσουμε προτεραιότητα αποζημίωση σε περίπτωση που ακυρώνεται κάποια υπηρεσία και να υπάρχει ε, ένα κατάλληλο έντυπο για υποβολή καταγγελιών και στο διαδίκτυο αλλά και ε, σε χειρόγραφο. Ε, εάν πραγματικά θέλουμε να αυξήσουμε τη χρήση των σιδηροδρόμων και πρέπει να εγγυηθούμε ότι έχουμε κατάλληλα ωράρια εργασίας, τα οποία να προσαρμόζονται και στα ωράρια εργασίας των επιβατών και να μην υπάρχουν αδικαιολόγητες και συχνές καθυστερήσεις, να υπάρχει προσοχή για τον πελάτη σε κάθε σταθμό. Και τέλος, ε, μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες με αυτή την έκθεση είναι ένα άλμα ποιότητας, ε, να υπάρχει πρόσβαση για τους ευάλωτες ομάδες. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία, συν άτομα τα οποία για λόγω ηλικία ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο μπορεί να έχουν μειωμένη κινητικότητα. Ε, όσοι χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται και να βοηθήσουμε ανθρώπους οι οποίοι σήμερα δεν μπορούν να μετακινηθούν τους πρέπει να έχουν ενημερώσει για να τους παρέχονται τα κατάλληλα μέσα. Η ε, ε, διαδικασία αυτή είναι φθηνή. Απλώς χρειαζόμαστε να αλλάξουμε λίγο όρομα. Να υπάρχει μια ράμπα, για παράδειγμα, στο τρένο, να μην υπάρχουν κλίμακες ε, και να διασφαλίσουμε ότι οι γραπτές πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες και από άλλους διάβλους. Πρέπει λοιπόν να δίνονται ε, τουλάχιστον οι ελάχιστες πληροφορίες ε, για τους φυσικούς ε, φραγμούς ε, και να μην υπάρχουν φραγμοί στην ενημέρωση για τους υπευθύνους και γι' αυτό ακριβώς είμαστε κατά της προειδοποίησης που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των 48 ώρων. Υπάρχουν παραδείγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αποδεικνύουν ότι αρκεί μία ώρα ή και χωρίς καμία προειδοποίηση. Είναι όλα θέλεμα διάθεσης, στρατηγικής και σωστή διαχείρισης. Ε, ε, μέτρα τα οποία μπορούν να δώσουν ε, δυνατότητα να βελτιώσουμε την ποιότητα με ελάχιστο κόστος και ελπίζουμε και την υποστήριξη των υπολείπων ομάδων στις τροπολογίες μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και έτσι ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις των σχεδόν εισηγητών. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που έχουν ζητήσει το λόγο. αν μπορούν να περιοριστούν στα δύο λεπτά Η κυρία Ρεβονταλόν έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπω έχω πει και προηγουμένω, η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κάτι το οποίο περιμένουν οι πολίτε για το θέμα αυτό, διότι είναι ε, άνοιγμα ε, για τον ανταγωνισμό για πολλά κράτη-μέλη. Ε, εδώ έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προστατεύει μόνο την απελευθέρωση των αγορών, αλλά και τα δικαιώματα των ε, επιβατών. Και διαβάζοντα τι τροπολογίε που υποβάλλονται, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε το κείμενο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιώσουμε τα δικαιώματα των επιβατών. Καταρχώς, ε, πολλοί ζήτησαν ε, ε, τροπολογίες για τις εξαιρέσεις των περιφερειακών αστικών και περιαστικών τρένων. Ε, καταλαβαίνω τις ανησυχίες πολλών συναδέλφων, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι περιφερειακές τουλάχιστον υπηρεσίες ε, εντάξει για τα αστικά και περιαστικά τρένα. Αλλά επίσης ε, δεν γίνεται να αποκλείουμε αυτές οι υπηρεσίες από τα δικαιώματα των επιβατών. Θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια μέχρι τέλους και να έχουμε άνοιχτα, άνοιγμα των δημοσίων υπηρεσιών αλλά και δικαιώματα δικαιώματα των επιβατών επί ίσης Το είπε και ο Μίχαλ Κράμερ. Ε, πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε μια λέση που επιτρέπει να λάβουμε υπόψη πολύ συγκεκριμένε περιπτώσει, όπω για παράδειγμα τη δυνατότητα να έχουμε και άλλα μέσα μεταφορά, αλλά δεν θα πρέπει ε, να διατηρήσουμε τον πιο αυστηρό ορισμό για την περίπτωση τη ανωτέρα βία. Και τέλος θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή του εισηγητή και των σχεδόν εισηγητών για τη δυνατότητα ε, στο δικαίωμα στην ανταπόκριση. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει το γεγονός ότι αυξάνονται οι επιβάτες που αλλάζουν μέσα μεταφορές ε, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σε μια διαδρομή. Ευχαριστώ. Η κυρία Άντερσον έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή που τόνισε το γεγονός ότι το θέμα αυτό είναι υψηλής ορατότητας και όπως υπόθηκε, εάν δεν προστατεύσουμε αποτελεσματικά τους επιβάτες με τις τροπολογίες μας και με το τελικό αποτέλεσμα, θα είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε στους ψηφοφόρους μας γιατί κάναμε αυτά που κάναμε. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η πολιτική μεταφορών και πάρα πολύ με ενδιαφέρει η συμμετοχή μου σε τούτη την Επιτροπή, αλλά θα γνωρίζετε ότι μερικές φορές θεωρείτε ότι η Επιτροπή μας δεν είναι υπέρ των ε, συμφερόντων, των ενδιαφερόντων των καταναλωτών. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω να σκεφτούμε προοδευτικά πάνω στο θέμα αυτό και θα ήθελα να ευχαριστήσω τις άλλες πολιτικές ομάδες για την ε, εξαιρετική συνεργασία. 106 τροπολογίες έχουμε υποβάλει εγώ και άλλοι συναδελφοί μου από την ομάδα S&D. Τι οποίε έχουν προσυπογράψει και βουλευτέ από άλλε πολιτικές ομάδες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία που είχε πολύ δύσκολη δουλειά με το θέμα αυτό, διότι πρόκειται για αναδιατύπωση και γι' αυτό είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο θέμα. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια θέματα. Ε, θα ήθελα να ε, επικροτήσω ιδιαίτερα αυτό που είπε ο κύριος Μιζελιέ για τις εξαιρέσεις. Ε, όλα τα στοιχεία της Επιτροπής δείχνουν ότι υπήρξε κατάχρηση των δυνατοτήτων εξαίρεσης από τα κράτη-μέλη και ε, ήρθε η ώρα να δούμε τη γενικότερη εικόνα και να τροποποιήσουμε ανάλογα τον κανονισμό αυτών. Θα ήθελα να στηρίξω επίσης ε, τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. το θέμα των κινητικών περιορισμών είναι κάτι το οποίο μπορούμε να λύσουμε χωρίς μεγάλες δυσκολίες ε, και δεν θα πρέπει να το αγνοήσουμε. Ιδιαίτερα στους μεγάλους ε, σταθμούς είναι εύκολο να γίνουν ρυθμίσεις ε, ώστε να βοηθηθούν τα άτομα αυτά. Επίσης θα ήθελα να ενισχύσουμε τους στόχους του κανονισμού αυτού, διότι θέλουμε να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των επιβατών και να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να πάρουν το τρένο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουν όλοι εδώ στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα επίσης να τονίσω τις τροπολογίες ε, για τις περιπτώσεις όπου χάνει κανείς ε, την ε, ανταπόκρισή του. Είναι σημαντικό να φτάνουν τελικά στον τελικό τους προορισμό οι άνθρωποι αυτοί και δεν είναι θέμα προαιρετική ε, προσέγγιση. Ε, ναι, κάποιε επιχειρήσει. Ε, λένε θα σα βοηθήσουμε, αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένη αξίωση, συγκεκριμένο δικαίωμα αν κάτι πάει στραβά. Και θα ήθελα να αναφέρω και την τροπολογία 355 τη Κριστίν. Και θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά που είδε είπε η Κριστίν. Όσον αφορά την ανωτέρα βία, καταλαβαίνω τη θέση του ECR, αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω να το σκεφτείτε προσεκτικά διότι είδαμε πάρα πολλές ε, δικαστικές υποθέσεις λόγω ανωτέρας βίας σε άλλες περιπτώσεις. Ε, ε, για παράδειγμα, σε περίπτωση απεργιών. Εγώ είμαι κατά αυτού, αλλά ήδη στο δικαστήριο την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε μια υπόθεση για την ανωτέρα βία σε περίπτωση προειδοποίητης απεργίας. Ε, είτε είναι νόμιμη είτε είναι παράνομη η απεργία, ε, είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τις ε, καλές εργασιακές σχέσεις. Δεν θέλουμε να καταλήξει στο δικαστήριο αυτή η νομοθεσία. Παρακαλώ ξανασκεφτείτε το θέμα της ανατερασβίας διότι δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο το θέμα αυτό. Η μελέτη αντικτύπου της Κομισιόν δείχνει ότι δεν θα ήταν σημαντικά τα ωφέλη για τις επιχειρήσεις. Παρακαλώ λοιπόν να το προσέξουμε πολύ προσεκτικά. Και επίσης θα ήθελα να εξυγχρονίσουμε τις ε, ρυθμίσεις. Ε, οι πράσινοι ανέφεραν ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι, αναφέ... ότι χρησιμοποιούμε περισσότερο ποδήλατα τα παραρτήματα του κανονισμού αυτού είναι τελείως παροχημένα. Μπορεί να διαφωνούμε όσον αφορά το επίπεδο ανάλυσης, αλλά θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το ε, αν υπάρχει δίκτυο Wi-Fi στο τρένο. Ακόμα και αν απλά λέμε δεν υπάρχει δίκτυο Wi-Fi. Είναι διατυπωμένα με πολύ παλιό τρόπο, ε, τα, ε, με παροχημένο τρόπο τα παραρτήματα. Και πιθανότατα το πιο σημαντικό θέμα εδώ είναι η επιβολή του νόμου. Πάρα πολλέ τροπολογίε έχουν υποβληθεί για τα άρθρα 28, 29, 32, 33 και 35. Διότι στην πράξη το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι ε, δεν μπορούν να ασκήσουν ε, οι άνθρωποι τα δικαιώματά τους. Ε, κάποιες συνδρομικές επιχειρήσεις τα καταφέρνουν καλά, κάποιες εθνικές αρχές τα καταφέρνουν καλά, αλλά σε άλλες περιπτώσεις όχι. Λυπάμαι που μακρηγόρησα, αλλά είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Κρασβάντα Ε, θα είμαι σχετικά σύντομη, διότι δεν θα επαναλάβω όλα όσα υπόθηκαν. Ωστόσο, ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κανονισμός αυτός. Ε, υπάρχουν κάποια σημεία παροχημένα τα οποία θα πρέπει να επανεξετάσουμε. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ελλείψεις και θα πρέπει να επικεντρωθούμε στους καταναλωτές, στους επιβάτες και να ενισχύσουμε τα δικαιώματά τους όσον αφορά το θέμα της ανωτέρας βίας. Δεν επιτρέπεται να φέρει ο επιβάτης τον κίνδυνο και όχι η επιχείρηση. Ο Μίκαελ Κράμερ είπε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των επιβατών στο θέμα αυτό, ώστε να μην ε, υπάρχουν ασάφειες. Όσον αφορά τους επιβάτες ε, με μειωμένη κινητικότητα. Υπάρχουν ε, ε, οι οι προθεσμίες για την προειδοποίηση σε μεγάλους σταθμούς όμως ε, δεν είναι απαραίτητη αυτή η εκ των προτέρων ειδοποίηση. Για να μπορέσει ο επιβάτης να πάρει το τρένο χρειάζεται η σχετική υποδομή καθώς και καταρτισμένο προσωπικό. Αλλά δεν θα έπρεπε αυτό να αποτελεί πρόβλημα. Σημαντικό είναι όλοι να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους σιδηροδρόμους, να γίνουν πιο ελκυστικοί και πιο φιλικοί προς το επιβάτη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Κουκασεύσκα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα μιλούμε για τα δικαιώματα των επιβατών στις σιδηροδρομικές μεταφορές και θέλουμε να προωθήσουμε τις σιδηροδρομικές μεταφορές, θέλουμε να δημιουργήσουμε κίνητρα, να παροτρύνουμε τους επιβάτες ε, να μεταφερθούν από τις οδικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Γιατί οι σιδηροδρομικές μεταφορές χρησιμοποιεί τρεις φορές λιγότερη ενέργεια από τις οδικές μεταφορές. Επίσης έχει λιγότερες ε, εκπομπές δημοσίου του θερμοκηπίου. Γι' αυτό θέλουμε να παρακινήσουμε τους ε, επιβάτες να χρησιμοποιούν περισσότερο τις ιδεροδρομικές μεταφορές. Και αν το καταφέρουμε, αν καταφέρουμε δηλαδή να θεσπίσουμε ένα κατάλληλο κανονισμό και για τους ιδεροδρομικές μεταφορές ε, ανάλογα με τις ε, αεροπορικές μεταφορές με αντίστοιχο δικαίωμα αποζημίωσης, πιστεύω ότι πραγματικά θα αυξήσουμε τη χρήση των σιδηροδρόμων. Γιατί αν δεν υπάρχει ευθύνη, αν δεν υπάρχουν συνέπειες, κανένας δεν θα καταβάλει τις προσπάθειες που χρειάζονται ε, για να ικανοποιήσει τους επιβάτες. Είμαστε στον 21ο αιώνα, οπότε θα πρέπει να έχουμε μία ενιαία ευρωπαϊκή πλατφόρμα, ώστε ο κάθε επιβάτης να μπορεί να βρίσκει ε, πληροφορίες για τα δρομολόγια και να αγοράζει ε, διαδικτυακά τα εισιτήριά του και μάλιστα να μπορεί να αγοράζει και ενιαίο εισιτήριο πολύ σωστά μιλήσαμε και για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα και αναπηρίες που θα πρέπει να έχουν ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπου ε, ε, υπόλοιπους ε, ε, επιβάτες και να μην πρέπει να προειδοποιεί εκ των προτέρων ο, το άτομο με μειωμένη κινητικότητα ότι θα χρειαστεί κάποια αρρωγή στο σιδηρόδρομο. Θα πρέπει να είναι εύκολη η παροχή τέτοια βοήθεια. Ελπίζω να ληφθούν υπόψη οι τροπολογίε μου, γιατί πραγματικά οι σιδηρόδρομοι είναι για τους επιβάτες. Χωρίς επιβάτες δεν θα έχουμε σιδηροδρομικές μεταφορές. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και κάποιοι συνάδελφοι που ε, φαίνεται ότι στέκονται στο πλευρό των επιχειρήσεων και όχι στο πλευρό των επιβατών ελπίζω ότι θα μεταπιστούν και θα... Ε, υποχωρήσουν κάπως τις προτάσεις τους, ώστε πραγματικά να κάνουμε επανάσταση και να μεταφέρουμε πολύ περισσότερους επιβάτες από τις οδικές μεταφορές στις σιδηροδρομικές. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ντεμόντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πρότασή του. Όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί ο στόχος αποτελεσματικών δικαιωμάτων για τους επιβάτες. Αλλιώς δεν θα ήμασταν εδώ να το συζητούμε μέχρι τώρα. Αλλά χρειαζόμαστε αυτή την αποτελεσματικότητα ακριβώς γι' αυτό το λόγο και η διάταξη είναι τόσο σημαντική. Εγώ έχω προσπογράψει κάποιες τροπολογίες, μεταξύ αυτών ε, η ουδετερότητα και η δυνατότητα να ε, συγκρίνει κάποιο ε, τι προσφορέ για να υπάρχει και πραγματική ανταγωνιστικότητα. Ε, ανταγωνιστικότητα η οποία δεν θα πρέπει να γίνεται μόνο όσον αφορά την τιμή, αλλά και όσον αφορά την ποιότητα τη υπηρεσία και επίσης μια τροπολογία όσον αφορά την πώληση ξεχωριστών εισιτηρίων. Διότι εγώ είμαι πεπισμένη ότι η ευθύνη για τις πληροφορίες δεν θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα της σιδηροδρομική υπηρεσίας, αλλά του πολιτή. Αυτή είναι μια γενική αρχή. Να υπάρχει δηλαδή μια διαμεσολάβηση και όταν υπάρχει διαμεσολάβηση θα πρέπει ο διαμεσολαβητή να παρέχει τι πληροφορίε και να είναι και υπεύθυνο γι' αυτό. Ε, άλλωστε αυτό να το σκεφτούμε γίνεται και στις πλατφόρμες. Πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στα άτομα με αναπηρία. Νομίζω ότι αυτό είναι το κεντρικό θέμα όταν συζητούμε για δικαιώματα επιβατών. Σε γενικές γραμμές ε, για τις πιο ευάλωτες κατηγορίες θα πρέπει να υπάρχει σίγουρα μια ρεαλιστική σχέση, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει και σαφήνεια και διάθεση να επιλύσουμε τα προβλήματα. Επομένως, ε, η πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς είναι ένα θέμα το οποίο εξακολουθεί να είναι κεντρικό ζήτημα και δεν έχει επιληθεί ε, τελικά. Ε, και αυτό αφορά και την καθημερινότητα ανθρώπων που καθημερινά πρέπει να μεταβούν στο χώρο της εργασίας τους, ακόμα και σε αυτούς όμως που χρησιμοποιούν περιστασιακά τα μέσα μεταφοράς, αλλά αυτό θα πρέπει να αφορά και την ανάπτυξη του τουρισμού, διότι μόνο το 4% των τουριστών ε, σήμερα χρησιμοποιεί μέσα μαζικής μεταφοράς ε, σε τοπικό επίπεδο. Όσον αφορά τη συνδρομή, θα πρέπει να να είναι εγγυημένη η αρρωγή χωρίς ε, να ε, υπάρχει πρόβλημα προστασίας προσωπικών δεδομένων, να παρέχεται δωρεάν και χωρίς διάκριση μεταξύ αστικών κέντρων και περιφερειακών κέντρων. Να υπενθυμίσω ότι η πρόσβαση δεν θα πρέπει να είναι μόνο η φυσική δυνατότητα πρόσβασης, που αυτό θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο, αλλά και πρόσβαση σε πληροφορίες, ε, πληροφορίες και εναλλακτικέ συνδέσεις. Ε, πολύ χάρηκα που άκουσα και από τους συναδέλφους σήμερα ε, τον ορισμό της ε, μεταφοράς για όλους, κινητικότητα για όλους. Επομένως η πρόσβαση δεν θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο εκχωρούμε, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι και εκτιμένο δικαίωμα για όλους τους επιβάτες. Η κινητικότητα θα πρέπει να εγγυάται σε όποιον έχει προβλήματα αναπηρίας, σε όποιον έχει προβλήματα προσωρινής κινητικότητας και θα πρέπει να λάβουμε και υπόψη ότι η κοινωνία μας γυράσκει. Επομένως ε, ε, ακόμα περισσότερο πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι θα πρέπει να τους διευκολύνουμε για να μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σας ευχαριστώ. Ο Δόκτωρ Κόρ έχει το λόγο τώρα. Κοχ, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την ε, πολύ καλή έκθεση του κυρίου Λιμπεράτσκι. Κάθε εβδομάδα ε, ε, ε, ε, κάνω μεγάλες διαδρομές με το τρένο για να έρθω εδώ στις Βρυξέλλες από την πατρίδα μου και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα για την αναδιατύπωση του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών. Κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά τους πολιτές των εισιτηρίων συμφωνώ με τον εισηγητή. Θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για το κλείσιμο του εισιτηρίου αλλά ε, ε, η συνδρομική επιχείρηση θα πρέπει να ενημερώνει αμέσως πριν το ταξίδι και κατά τη διάρκεια του και όχι ένας ανεξάρτητος ε, ταξιδιωτικός πράκτορας. Πληροφορίες πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αυτό δεν είναι δύσκολο στις μέρες μας με την τεχνολογία που υπάρχει στη διάθεσή μας. Τρίτον, τα through tickets. Ούτε και αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν πρόβλημα. Δεν ε, θα ήθελα να πρέπει να εξηγήσω σε έναν Ευρωπαίο ε, που θέλει να πάρει το τρένο από τη Βαϊμάρη στο Παρίσι γιατί δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους οι συνδρομικές επιχειρήσεις. Ε, δεν θα πρέπει να ανήκουν στο μέλλον αυτά τα ενιαία στήρια, θα έπρεπε ήδη να τα έχουμε εισάγει. Όσον αφορά το να μπορεί να παίρνει κανείς μαζί του το ποδήλατο, αυτό είναι, πάρα πολύ... αυτό είναι απολύτως απαραίτητο και για τους εργαζόμενους και για τον τουρισμό. Γι' αυτό στην τροπολογία μου ε, θέλω οι δυνατότητες παρέκκλησης ε, να περιοριστούν. Και πέμπτον, το πιο σημαντικό θέμα και για μένα είναι τα δικαιώματα των ε, ανθρώπων με μειωμένη κινητικότητα. Γνωρίζω το Ολλανδικό μοντέλο που παρέχει βοήθεια με προειδοποίηση μιας ώρας. Ξέρω ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει σε όλες τις άλλες χώρες και σε κάθε μικρό σταθμό. Ωστόσο, θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τους μεγάλους συνδρομικούς σταθμούς. Και έχω υποβάλει σχετική την οποία ελπίζω να υπερψηφίσετε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν ε, ε, με τις παρεμβάσεις των συναδέλφων να δώσω το λόγο στον κύριο Ολιβιέ Νέρ από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μας πει την άποψη της Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει το μεγάλο ενδιαφέρον που έχουν δείξει τα μέλη της Επιτροπής σας ε, για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δικαιώματα των ε, επιβατών των σιδηροδρόμων. Πολλές από τις 637 τροπολογίες που έχουν προταθεί μέχρι τώρα θέλουν να διευκρινίσουν περαιτέρω τα δικαιώματα των επιβατών, να, αυξήσουν την, να αυξήσουν συγγνώμη, την ασφάλεια δικαίου που είναι πολύ σημαντικό και να επιτύχουν μια καλή συμφωνία μεταξύ ρεαλισμού και φιλοδοξίας. Επομένως σας ευχαριστώ. Ωστόσο, Ταυτόχρονα, κάποιες από τις προτινόμενες τροπολογίες ξεφεύγουν από τους στόχους της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι η βελτίωση της εφαρμογής των δικαιωμάτων των επιβατών και να διασφαλίσουμε ότι ε, θα μπορούν να λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα των επιβατών και να υπάρχει προστασία του τομία και έμεσα και ε, προστασία των επιβατών. Ε, νομίζω λοιπόν ότι σε αυτό το στάδιο της συζήτησης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υπενθυμίσει απλώς ε, κάποιες ε, βασικές εξελίξεις οι οποίες προτείνονται στο κείμενό μας, όπως για παράδειγμα η άρση των εξαιρέσεων που υπάρχουν για τις ε, χώρες υπηρεσίες, καλύτερη ενημέρωση των επιβατών όσον αφορά τον τύπο των προϊόντων που ε, παρέχονται, περιορισμένο πεδίο εφαρμογή της ανωτέρας βίας, κάτι το οποίο συζητήθηκε και σήμερα το πρωί, και επίσης ενίσχυση ε, των δικαιωμάτων των επιβατών με αναπηρία. Ευχαριστώ. Οπότε, πριν ολοκληρώσουμε, θα δώσουμε και πάλι το λόγο στον εισηγητή μας, τον Μπογκούσαφ Λιμπεράτσκι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους αξιότιμους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους. Κάθε συνάντηση και κάθε συνεδρίαση με γεμίζει με μεγαλύτερη ισοδοξία για την έκβαση. Γιατί Φαίνεται ότι συγκλίνουμε όλο και περισσότερο και προσβλέπω σε αίσιο πέρα τη διαδικασία. Βασικέ ε, ιδέε και βασικά ζητήματα. Τα είπε η κυρία Ντεμόντε. Προσβασιμότητα. Θέλουμε προσβάσιμους σιδηροδρόμους σε όσο το δυνατό περισσότερους επιβάτες. Δεύτερον, ελκυστικότητα. Ως προς τις τιμές, να είναι προσιτές οι τιμές. Ε, ως προς τις ε, συμπληρωματικές υπηρεσίες, ε, της την άνεση. Η ιδέα μου είναι να επιτρέψουμε στους επιβάτες να ξανανακαλύψουν τους σιδηροδρόμους. Και θέλουμε έναν ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο που δεν θα περιορίζεται στα εθνικά σύνορα. Θέλουμε έναν ενίο ανοιχτό ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο που μπορεί να καλύπτει όλες τις ε, μορφές και κατηγορίες ε, των υπηρεσιών προς τους ε, επιβάτες. Αστικές, προαστιακές, περιφερειακές, ναι. Ε, νομίζω ότι ως προς αυτό αρχίζουμε και συγκλίνουμε. Ε, Ευχαριστώ τους κύριους Μιζελίε, Πορέμπα, Κράμερ, τους παρόντες και οδησηγητές που παρουσίασαν με ξεκάθαρο τρόπο τις απόψεις τους. Οπότε, δεν νομίζω ότι υπάρχουν παρεξηγήσεις, γι' αυτό και θα επικεντρωθώ σε, στα βασικά σημεία για να συνεννόμαστε. Πεδίο εφαρμογή. Σε ποιο βαθμό θα εφαρμόσουμε τον κανονισμό. Δεύτερον, πληροφορίες ε, προς τους επιβάτες ε, τρίτον, ε, ποδήλατα ε, που μπορούν να επιβάζονται στα, στους σιδηροδρόμους, εξαιρέσεις, εισιτήριο, προσβασιμότητα των ατόμων με ε, μειωμένη κινητικότητα και αναπηρίες, ε, αποζημίωση και καθυστέρηση, ε, περιπτώσεις και καθυστερήσεων, το θέμα της ανωτέρας βίας και τι εμβέλεια θα έχει. Γιατί αρχικά υπήρχε μεγάλη διάσταση απόψε μεταξύ αυτών που απέρριπταν τελείω την ανωτέρα βία και αυτών που ήθελαν διασταλτική ερμηνεία τη ανωτέρα βία. Τώρα δεν την απορρίπτει κανένα. Το θέμα είναι τι θα περιλαμβάνει η ανωτέρα βία. Θα περιλαμβάνει και τι απεργίε. Ε, θα περιλαμβάνει και σεισμούς για παράδειγμα κατά τη γνώμη μου, στις, το θέμα των διαπεριφερειακών και των εθνικών σιδηροδρόμων εξετάζεται και θα ήθελε οι σιδηροδρόμοι να μπουν και πάλι ε, να είναι πάλι ανταγωνιστικοί σε σχέση με κάποιους μεταφορείς ε, χαμηλών, χαμηλού κόστους, του low cost. Εγώ μένω στη Βαρσοβία, 600 χιλιόμετρα μακριά και την περασμένη Κυριακή στις 7 το απόγευμα το τελευταίο, ε, το τελευταίο λεωφορείο ε, low cost, Λονδίνος Τσέτσιν, σε 50 λεπτά ε, σε πάει στο αεροδρόμιο και 180 ήταν οι επιβάτες, ενώ ε, τα τρένα μας κυκλοφορούν μισοάδια. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ανταγωνιστικές τις σιδηροδρομικές μεταφορές με, ισότιμες, όρους, με ισότιμους όρους ανταγωνισμού με τους μεταφορείς low cost για να κερδίσουμε το παιχνίδι του ανταγωνισμού χάρη των σιδηροδρόμων μας. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, ευχαριστώ για τις προτάσεις σας και τώρα περνάμε στην επόμενη φάση, στην κατάρτιση δηλαδή των συμβαστικών τροπολογιών και στη συνέχεια στην κατάρτιση του καταλόγου ψηφοφορίας. Σας ευχαριστώ, ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Οπότε ολοκληρώνουμε τη συζήτηση για αυτό το σημαντικό θέμα. Να σας υπενθυμίσω ότι η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα γίνει στις 21 Ιουνίου τρέχοντος έτους. Ε, το επόμενο σημείο της ημερήσης διάταξης θα συζητηθεί και κλεισμένο το θύρον. Γι' αυτό να αποχαιρετήσω όσους οφείλουν να αποχωρήσουν για αυτό το τμήμα της συνεδρίασης, γιατί θα έχουμε επαναλαμβάνω, και κλεισμένο το θηρό να κρώσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα πεντάλεπτο διακοπή για να κοινωθεί αίθουσα από όσου δεν δικαιούνται να είναι μέσα.